Okay. Good morning. Καλημέρα σας. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης τροποποίηση του κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και μελέτη των ε, τροπολογιών και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή Λεωνάρδο Ντομένιτσι. Ντομενίτσι, ε, μιλήτρια στην αρχή, το διόρθωσε Ντομενίτσι. Κυρία Πρόεδρε, μόνο δύο σκιώδεις εισηγητές βρίσκονται εδώ, κυρία Πρόεδρε. Μήπως θα μπορούσαμε να περιμένουμε τουλάχιστον τον κύριο Κόζες. Ε, βρίσκεται σε μια συνεδρίαση, λέει η Πρόεδρος, και μας είπε να ξεκινήσουμε χωρίς αυτόν. Δεν έχουμε το ΕΛΚ, έχουμε το ΑΛΔΕ. Ο Φελίπ νομίζω θα μιλήσει για τον Κασκάου. Έχουμε λοιπόν τρεις ομάδες έτοιμες και έτσι θα μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς αυτόν όπως με ζήτησε. Ωραία λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε κάμποσο χρόνο στη διάθεσή μας για αυτή τη συζήτηση. Ίσως να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε όλο, αλλά αναμένοντας μέχρι να φτάσουν οι άλλοι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Στο μεταξύ, ως πρώτη παρατήρηση θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και και τους συναδέλφους της Κομισιόν που συνέβαλαν ο καθένας με τον τρόπο του σε αυτή την έκθεση με την παρουσίαση μιας, ε, ενός αρκετά μεγάλου πλήθους τροπολογιών και ελπίζω ότι μετά από τη συζήτηση σήμερα το πρωί θα μπορέσουμε να εργαστούμε επικοδομητικά ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες θα αποτυπώνουν ε, τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ορισμό αυτού του νέου κανονισμού. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, διαιρώντας, διχωρίζοντα τα επιχειρήματα σε δύο κατηγορίες. Αναγνωρίζονται βάσει των τροπολογιών έξι ζητήματα, έξι ερωτήματα. Ενδεχομένως θα προσθεθούν άλλα κατά τη διάρκεια της συζήτησης και έτσι θα μπορούσαμε να τα εμβαθύνουμε τρία ζητήματα που θεωρώ ύψης της σημασίας. Φυσικά αντιφατικά ζητήματα και που προκαλούν κάποια προβλήματα αφορούν την ε, εναλλαγή, την ε, πιστοληπτική αξιολόγηση των ε, κρατικών χρεών και την κοινωνική ευθύνη. Και επίσης άλλα τρία επιχειρήματα τα οποία με τα οποία θα ασχοληθώ στη συνέχεια. Η μεθοδολογία over alliance και η σύγκρουση ε, συμφερόντων για τα οποία θεωρώ ότι θα είναι πιο εύκολο να επιτύχουμε κάποια σύγκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσω μιλώντας ε, χωρίς ε, γενικές περιστροφές για το ζήτημα των κρατικών χρεών, των δημοσίων χρεών. Θεωρώ ότι αυτός ο νέος κανονισμός έχει νόημα και μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός εφόσον εμείς δώσουμε μια απάντηση και αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και το ζήτημα της ε, αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ε, των κρατομελών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επ' αυτού θα ήθελα, αν μου επιτρέπουν ε, οι συνάδελφοι, να πω δυο λόγια για την πρόταση που παρουσιάστηκε από εμένα ως εισηγητή απαγόρευσης των unsolicited ratings, ε, δηλαδή των ε, αξιολογήσεων χωρίς να έχουν ζητηθεί για τα κρατικά χρέη. Ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι και αυτό προέκυψε με τη, στη συνεδρίαση με το ΣΕΝΤΟΣ ε, εξέφρασαν προβληματισμούς όσον αφορά αυτή την πρόταση. Οι οποίοι προβληματισμοί είναι απολύτως εύλογοι. Ωστόσο, εγώ θα επιθυμούσα να εξηγήσω κάπως καλύτερα ποιο είναι το σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται αυτή η πρόταση. Όχι με στόχο να επιμείνω απλά για την επιμονή, αλλά για να δώσουμε νόημα σε αυτή την κοινή έρευνα, αναζήτηση, επιδίωξη που κάνουμε για να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Η πιστοληπτική αξιολόγηση του κρατικού χρέου, του δημοσίου χρέους, έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάποια ιδιαιτερότητα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον προβληματισμό μας. Οι επιπτώσεις μιας αξιολόγησης δημοσίων χρεών δεν είναι οι ίδιες επιπτώσεις με εκείνες μιας, ενός άλλου τύπου αξιολόγησης. Γι' αυτό το λόγο απαιτείται κατά την άποψή μου ε, ιδιαίτερο κανονιστικό πλαίσιο. Η πρόταση απαγόρευσης του unsolicited rating για τα δημόσια χρέη θα πρέπει να συσχετιστεί με την άλλη πρόταση την πρόταση θέσπισης ε, ενός δημόσιου ανεξάρτητου οργανισμού ο οποίος ε, θα επιτελεί το καθήκον ε, εκτέλεσης της αξιολόγησης των δημοσίων χρεών. Ορισμένοι συνάδελφοι έφεραν αντίρρηση λόγω του ότι υπάρχει περίπτωση να περιορίζονται οι δράσεις αξιολόγησης λόγω αυτής της απαγόρευσης. Θεωρώ ότι αυτή η σκέψη είναι σημαντική. Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν είναι απολύτως βάσιμη. Εξαιτία των όσων είπα προηγουμένως, των ιδιαιρωτήτων, των επιπτώσεων των αξιολογήσεων πιστοληπτικών ικανοτήτων για τα δημόσια χρέη το γεγονός ότι το επιχείρημα που αφορά την ελευθερία μπορεί να ανατραπεί διότι ε, με αυτόν τον τρόπο θα έχει ένα κυρίαρχο κράτος την ελευθερία να επιλέξει κατά πόσο θα αξιολογείται από ιδιωτικές εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή κατά πόσο θα ε, επαφείται αποκλειστικά σε μία αυτόνομη και ανεξάρτητη οντότητα. Θεωρώ ότι το σημείο αυτό είναι σημαντικό. διότι ούτως ή άλλως οι πληροφορίες ε, θα παρέχονταν στους επενδυτές από αυτό τον αυτόνομο και ανεξάρτητο οργανισμό όσον αφορά το δημόσιο χρέος και οι επενδυτές ούτως ή άλλως θα έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε μια εταιρεία αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτική, ώστε να ζητήσουν μια αξιολόγηση, μια αξιολόγηση από εκεί και όσον αφορά τα δημόσια χρέη. Φυσικά αυτό το σημείο θα πρέπει να μελετηθεί και υπό μια άλλη πτυχή κατά την απόψή μου, πράγματι το ενδεχόμενο απόρριψης αυτής της ε, απαγόρευσης αξιολόγησης των δημόσιων χρεών ε, δεν αποκλείει την πρόταση δημιουργίας ε, ενός θεσμού που θα πραγματοποιεί τέτοιες αξιολογήσεις ανεξάρτητα και αυτόνομα στο πλαίσιο των υπαρχόντων ευρωπαϊκών οργάνων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων που θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση των δημοσίων χρεών της ε, πιστοληπτικής ουσιαστικά ικανότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επ' αυτού θεωρώ την ενδιαφέρουσα τροπολογία που παρουσιάστηκε από τον συνάδελφο Φέιο, τροπολογία 380, με τίτλο «Αρχή Ευρωπαϊκή για το χρέος» Ευρωπαϊκή Αρχή για το Χρέος που πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση με τα όσα πρότεινα εγώ. Η αρχή που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά και στην περίπτωση της αξιολόγησης της πιτροληπτικής ικανότητας ε, των ε, δημοσίων χρεών. Η αρχή λοιπόν αυτή είναι ότι υπάρχει πολυφωνία και δυνατότητα σύγκρισης αυτών των διαφορών απόψεων οδηγούν σε μεγαλύτερη αξιοπιστία των αξιολογήσεων. Και αυτό ισχύει ως αρχή τόσο στον ε, δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό. Όσον αφορά αυτή την πτυχή της ε, δημιουργίας μιας οντότητας με αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να επιτελεί αυτό το ρόλο, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο άμεσα ή έμεσα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το επιχείρημα αποτέλεσε το αντικείμενο μια συνάντηση που είχα χθε μετά από τον νομισματικό διάλογο με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μάριο Ντράγκη, κατά την οποία συζήτηση δεσμεύτηκε να αξιολογήσει και να εμβαθύνει το ερώτημα και να δώσει σε εμάς, σε και μέσω στο κοινοβούλιο μια απάντηση εντό το πολύ τριών εβδομάδων. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα και όσον αφορά την κεντρική τράπεζα και γενικότερα το σύστημα κεντρικών τραπεζών υπάρχει ήδη σημαντική τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των δημοσίων χρεών που υπάρχει στο πλαίσιο του ECAF, του Euro System Credit Assessment Framework, στο το οποίο αναφέρεται και σε κάποιες από τις τροπολογίες που παρουσιάστηκαν. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ εγώ ότι η δυνατότητα χρήσης της τεχνογνωσίας που ήδη υπάρχει μέσω των κεντρικών ας πούμε, εθνικών τραπεζών θα μπορούσε να επιφέρει Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζονται και από πολλέ τροπολογίε, θα μπορούσε λοιπόν να οδηγήσει τους, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αναπτύξουν ίδια συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγηση, όπω εξάλλου ζητείται από πολλέ τροπολογίε. Ε, αναφέρω για παράδειγμα τι τροπολογίε του συναδέλφου Καμφά, ε, αλλά υπάρχουν και πολλέ άλλε. Πιστεύω ότι η πολυφωνία θα μπορούσε να έχει επίσης ως συνέπεια να μετριάσει το προκυκλικό φαινόμενο τις προκυκλικές επιπτώσεις ορισμένων αξιολογήσεων όπως έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν για τα δημόσια χρέη. Επ' αυτού θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τη συνεισφορά εφόσον υποθέσουμε ότι θα υπάρξει κάποιο συμβιβασμός που θα προέλθει από κάποιες τροπολογίες όπως των συναδέλφων Κλίντς και Γκοζές αλλά και Ασλεφόξ που σχετίζονται με τη δυνατότητα ενός προληπτικού χρονοδιαγράμματος ή ε, κατά κάποιο τρόπο ε, κάποιων χρονικών ε, καθορισμών των αξιολογήσεων. Αυτά ως ε, αφετηρία για την αξιολόγηση των δημοσίων χρεών προσπάθησα να σας εξηγήσω και να επιχειρηματολογήσω όσο γίνεται καλύτερα για την άποψή μου αλλά θεωρώ ότι οι τροπολογίες που ανέφερα αποτελούν και σημαντικές συνεισφορές ώστε να μπορέσουμε να επιδιώξουμε ε, προηγμένου επίπεδου συμβιβασμούς. Περνάω στο δεύτερο σημείο, το οποίο αποτελεί ίσως την πιο αντιφατική και προβληματική ίσως πτυχή για την οποία έχει γίνει πολλές συζητήσεις. Αυτό που έχει σχέση με την εναλλαγή. Ορισμένοι συνάδελφοι προτείνουν την κατάργηση της ακύρωσης που προτείνεται από την Κομισιόν για την ε, περιοδική εναλλαγή των ε, οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Εγώ συμφωνώ ότι η διατύπωση που περιλαμβάνεται στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής ενέχει πτυχές περίπλοκες όσον αφορά την εφαρμογή Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε το καθήκον να πραγματοποιήσουμε μια προσπάθεια για να καταδείξουμε πιθανές λύσεις εναλλακτικέ βάσει της βασικής αρχής, της θεμελιώδους αρχής που εμπνέει αυτή την πρόταση της Κομισιόν. Ήτι ένα μέγιστο ανοίγμα της αγοράς περισσότερες δυνατές ε, ε, περιπτώσεις ανταγωνισμού, οι μεγαλύτερες δυνατές δυνατότητες ανταγωνισμού. Κατά την απόψή μου λοιπόν έχουμε δύο πιθανές οδούς μπροστά μας. Η πρώτη είναι εκείνη που προτείνουν ορισμένοι συνάδελφοι Σκέφτομαι, τώρα έχω στο νου μου τις τροπολογίες της κυρίας Μπόλς, του Καμφά, του Τόμας Μάν, αλλά και τις προτάσεις που προήλθαν ε, ε, παρότι από το Συμβούλιο. Η πρώτη οδός λοιπόν είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την περιοδικότητα της εναλλαγής ε, βάσει συγκεκριμένων προβληματισμών, συγκεκριμένων προϋποθέσεων ή αλλιώς πάντα στο ίδιο πλαίσιο και ε, στα κριτήρια που προτείνονται από τους Κλούντε και Κώστας που ήθελα να επιθυμίσω όσον αφορά τα όρια συγκέντρωσης ε, πλήθους αξιολογήσεων ανά ε, εκδότη. Αυτή είναι η πρώτη οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε με βάση το γεγονός ότι ούτως ή άλλως που ούτως ή άλλως η Κομισιόν προτείνει με τον νέο κανονισμό. Η δεύτερη εναλλακτική είναι να δουλέψουμε για ένα εναλλακτικό σύστημα το οποίο θα διατηρεί όπως έλεγα προηγουμένως τον απότερο σκοπό της εναλλαγής μέσω συνδυασμού προτάσεων. Έχω στο νόμο την τροπολογία 264 του κ. Γκόζες όπου εισαγάγει τη δυνατότητα μιας ε, ενός ε, δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή των οργανισμών αξιολόγησης πιστολοπτικής ε, ικανότητας. Την, σκέφτομαι την τροπολογία 265 της Ashley Fox για την εγγύηση της, του ανταγωνισμού, την τροπολογία 268 του Wolf Klintz σε σχέση με τους εκδότες που έχουν υποστεί αξιολόγηση και τη δυνατότητα ε, εισόδου των μικρών οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Χρειαζόμαστε ωστόσο έναν πιο ακριβή ορισμό του τι είναι Small Credit Rating Agency. Υπό αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο, πρόκειται εδώ για μια υπόθεση δική μου την οποία θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε καλύτερα στο μέλλον, της εισαγωγής μιας ε, υποχρέωσης άνω των δύο αξιολογήσεων ανά εταιρεία. Αυτές είναι οι δύο οδοί που έχουμε μπροστά μας. Από τη μία δουλεύουμε πάνω στο σύστημα που προτείνει η Κομισιόν με τις τροπολογίες, τροποποίησεις που προτείνουν ορισμένοι συνάδελφοι. Αφετέρου μπορούμε να προωθήσουμε εναλλακτικέ λύσεις που ωστόσο θα διατηρούν αυτό τον απότερο σκοπό ανοίγματο της αγοράς ε, του ανταγωνισμού που όπως υπενθύμησα ε, προηγουμένως αποτελεί το αντικείμενο των τροπολογιών άλλων συναδέλφων. Περνάω στο τρίτο σημείο που είναι πιο περίπλοκο και πιο αντιφατικό. Σχετίζεται με την εισαγωγή της αρχής της αστικής ευθύνης, civil liability για τους οργανισμούς αξιολογής πιστοληπτικής ικανότητας. Και σε αυτή την περίπτωση ορισμένοι συνάδελφοι προτείνουν να αποθήσουμε την αρχή της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης εις βάρος των εταιριών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Και σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να συστήσω μεγάλη προσοχή. Διότι θεωρώ ότι παρότι είναι συζητήσιμη, αυτή η πρόταση αντιστροφής ε, του βάρους της απόδειξης βασίζεται σε μία αρχή και σε μία βασική έννοια που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή, στο γεγονός ότι εμείς πρέπει να θεωρούμε εκ των προτέρων ότι υπάρχει μία ασυμμετρία των πληροφοριών μεταξύ του επενδυτή και του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που μπορεί να δικαιολογήσει σε περίπτωση αγωγής κατά της, ε, του οργανισμού αξιολόγησης ε, την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης και να θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή η πρόταση γενικά επιτελεί μια αποτρεπτική ουσιαστικά λειτουργία όσον αφορά τη λειτουργία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Φυσικά αυτό με αυτό δεν έχω πρόθεση να πω ότι η πρόταση πρέπει να παραμείνει ως έχει. Θεωρώ μάλιστα ότι πρέπει να αναλυθεί και να διερθρωθεί καλύτερα, διατηρώντας ωστόσο και εδώ αυτή την αρχή. Θεωρώ για παράδειγμα ότι θα μπορούσαμε να εισάγουμε μία αρχή βάσει της οποίας ο Οργανισμός Αξιολογικής Πιστοληπτικής Ικανότητας σε περίπτωση ε, μιας σοβαρής παράληψης ή μάλλον ε, πραγματοποιεί σοβαρή παράληψη αν παραβιάσει μία από τις προϋποθέσεις του παραρτήματος 3 του νέου κανονισμού ή σε περίπτωση παραβίασης γενικών υποχρεώσεων πίστης και επιμέλειας εκτός αν αποδείξει ότι αυτό αποτελεί ελαφρύ σφάλμα. Ζητώ συγγνώμη, εδώ τώρα ο τομέα είναι πιο νομικός και ε, χρειαζόμαστε αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, διότι και η ορολογία είναι λίγο πιο νομική. Ε, θα μπορούσε να μας δώσει κάποια εμβαθύνση η Επιτροπή Γιούρη. Η άλλη πτυχή είναι ότι μπορούμε να εγκαταλείψουμε αυτή την αρχή, να αφήσουμε αυτή την αρχή, συγγνώμη, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο επενδυτής θα πρέπει να παρουσιάζει με επαρκείς λεπτομέρειες με επαρκή επιμέλεια, με ε, σοβαρούς δείκτες από τους οποίους μπορούμε να συνάγουμε ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έχει πραγματοποιήσει μία από τις σοβαρές παραβιάσεις για τις οποίες μίλησα προηγουμένως. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι είναι σωστό ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να πρέπει να αποδείξει ότι έχει αναλύσει επιμελώς όλες τις σχετικές πληροφορίες, τις πληροφορίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας βάσει της κατάλληλης μεθοδολογίας και θεωρώ επίσης ότι ούτως ή άλλως εδώ το θέμα είναι να μπορεί να αποδείξει ότι οι πληροφορίες προέρχονταν ούτως ή άλλως από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές. Υπογραμμίζω αυτό το σημείο. Κυρίως αυτό το τελευταίο σημείο που αφορά την απόδειξη εκ μέρους του οργανισμού αξιολόγησης της αξιοπιστίας ε, των εργασιών της, διότι κατά την άποψή μου αυτό θα ευθυγράμμιζε τη δική μας πρόταση με τον Dodd-Frank Act, που θεωρώ είναι μια πτυχή σημαντική που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Μαζί με αυτό θεωρώ εγώ ότι η πρόταση για την αστική ευθύνη θα μπορούσε και να περιγραφεί πιο λεπτομερώς και να ενισχυθεί εισάγοντας πρώτα απ' όλα την, μια πλέον καθαρή, μια πιο καθαρή αρχή εναρμόνισης των δικαιοδοσιών δηλαδή το πιο δίκαιο ισχύει και σε πιο δίκαιο μπορεί να έχει κανείς προσφυγή από τη δική του χώρα δηλαδή σε πιο δίκαιο είναι εγγεγραμμένοι οι τίτλοι τη στιγμή της αγοράς. Δεύτερον, η ανάγκη πιο σαφής, σαφούς σχέσης μεταξύ της εποπτικής αρχής και των εθνικών δικαστικών αρχών και αυτό είναι πολύ σημαντικό κυρίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Τρίτον, την εισαγωγή μιας αρχής αναλογικής ευθύνης. Δηλαδή να γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών περιπτώσεων, δηλαδή το, η πραγματική εμβέλεια της ζημίας, τη διάκριση μεταξύ ενός θεσμικού και μη θεσμικού επενδύτη, ε, το ενδεχόμενο σφάλμα του ενδιάμεσου επενδυτή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα θέματα αστικής ευθύνης και την πρόταση μη απόρριψης της ε, δυνατότητας αντιστροφής ε, του βάρους της απόδειξης αλλά μπορούμε να καθορίσουμε πιο λεπτομερώς διευκρινίζοντας ορισμένες πτυχές την εφαρμογή αυτής της αρχής. Τώρα θα, έρθω, θα μιλήσω λίγο πιο γρήγορα για τα άλλα τρία σημεία τα οποία, ε, στα οποία αναφέρθηκα και τα οποία αφορούν το over Alliance τη μεθοδολογία και τη σύγκρουση συμφερόντων. Θα είμαι πιο γρήγορο γιατί θεωρώ ότι σε αυτά τα τρία σημεία οι δυνατότητες σύγκληση και συμφωνίας είναι πολύ μεγαλύτερε. και δεδομένης της τρέχουσας κατάσταση των πραγμάτων θα είναι πιο εύκολο να καταλήξουμε σε ε, σύγκληση. Ειδικότερα όσον αφορά το over Alliance Νομίζω ότι κατά βάθο ε, συμφωνούμε όλοι για τις αρχές και του στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν. Θα προτείνω να λάβουμε υπόψη την τροπολογία αριθμό 4 ε, του paper που περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με το over-alliance, με την υπέρμετρη δηλαδή εξάρτηση από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, που πιστεύω περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προτάσεις. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να μελετήσουμε το ενδεχόμενο προσέγγισης της μεταβατικής περίοδου για την υλοποίηση αυτής της αρχής ε, της ε, μείωσης της υπερβολικής εξάρτησης μέσω της αναθεώρησης της νομοθεσίας και των ισχυρών των κανονισμών. Εγώ πρότεινα διάστημα 6 μηνών. Ο κύριος Γκοζές πρότεινε τρία χρόνια. Πιστεύω ότι σε αυτού θα μπορέσουμε να συγκλίνουμε κατά κάποιο τρόπο. Υπογραμμίζω ωστόσο ότι όσον αφορά την υπέρμετρη εξάρτηση, το γεγονός ότι γίνεται αυτή η συζήτηση για το ρόλο και τη λειτουργία των οργανισμών εξολευσής πιστοληπτικής κανότητας ήδη επιφέρει σε ορισμένες περιπτώσεις μια νέα διάσταση όσον αφορά την εμπιστοσύνη που δείχνει το κοινό, οι βιομηχανίες, ε, οι πιστοτικοί οργανισμοί σε αυτούς τους οργανισμούς εξολέξης πιστοληπτικής ικανότητας όπως στη Δανία που θεωρώ δεν είναι αρνητικό. Όχι για λόγους τιμωρίας, των οργανισμών αξιολόγησης αλλά για την ανάπτυξη μιας, ε, εκείνης της πιο πολύπλοκης αυτονομίας της αξιολόγησης κυρίως εκ μέρους των επενδυτών στην οποία θα βασιστεί και θα, από την οποία θα εμπνευστεί ο νέος κανονισμός. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, και αυτό είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό. Και έχουμε να μελετήσουμε πολλά γι' αυτό και όσον αφορά τη διαφάνεια των μεθόδων και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι ιδιαίτερα ευρεία, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, ε, είναι πρόσφατο αυτό το γεγονός. Ε, η πρόσφατη αναγγελία υποβάθμισης ορισμένων τραπεζών στις Ηνωμένε Πολιτείε οδήγησε σε μια αρκετά στεναρή ε, πολεμική μάχη ουσιαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το κατά πόσο είναι αξιόπιστα ορισμένα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση αυτής της ε, υποβάθμισης. Εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά τη μεθοδολογία υπάρχει δυνατότητα να βρούμε ένα σημείο σύγκλησης. Διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο ρόλος του Τη ΕΣΜΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών θα πρέπει να είναι ρόλος επαλήθευση ελέγχου, αλλά ότι δεν έχει στόχο να δίνει κάποια σήμα ποιότητας. Πιστεύω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Αυτό που υπογραμμίζουν ορισμένοι συνάδελφοι, θυμάμαι καλά ο κύριος Γκοζές κυρίως, ε, θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να θα συμφωνήσουμε σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Χρειάζεται διευκρίνηση ορισμένα σημεία, αλλά γενικά συμφωνούμε όσον αφορά ε, αυτό το σήμα ε, αξιολόγησης της ΕΣΜΑ. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστούν ορισμένες τροπολογίες ε, οι οποίες, με τις οποίες προτείνεται η ανάγκη, η καταλληλότητα να ληφθούν υπόψη ορισμένα συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να εισαχθούν στην έκδοση αξιολογήσεων. Αναφέρομαι στην τροπολογία Κανφέν που σχετίζεται με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις ε, τροπολογίες Πλούτεν και Καμφά που σχετίζονται με την εισαγωγή και τη χρήση της, ε, ε, της πιθανότητας default. Τέλος, το τελευταίο κομμάτι όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων και εδώ πιστεύω είναι δυνατόν να εργαστούμε με τρόπο, να συνεργαστούμε θετικά, διότι οι τροπολογίες τείνουν να συγκλίνουν όσον αφορά τη διαφάνεια, όσον αφορά το πρόβλημα της υπέρβασης ε, όλων των κατοφλίων όσον αφορά τι διασταυρούμενε μετοχικέ συμμετοχέ. Ε, η αρχική πρόταση της Κομισιόν ήταν ε, ένα κατόφλιο του 5% και ξεκινώντας από μια δική μου τροπολογία, τον αριθμό 29, ενδεχομένω θα έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό όσον αφορά τα δελτία συγχώνευση που είχε προαναγγελθεί ούτω ή άλλως από τον Επίτροπο Μπαρνιέ πριν από την επίσημη παρουσίαση του νεοκανονισμού. Ωστόσο, στη συνέχεια ε, παραλήφθηκε πριν από την επίσημη παρουσίαση του ίδιου του κανονισμού. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη για όλο το χρόνο για τον οποίο μίλησα. Η παρουσίασή μου ίσως να περιέχει κάποια κενά, κάποιες ελλείψεις και είμαι βέβαιος ότι εσείς θα μπορέσετε να απαντήσετε θετικά ε, συμπληρώνοντας με τη δική σας συνεισφορά, με, τις ε, με τα δικά σας σχόλια. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια σκέψη γενικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι το ζήτημα των οργανισμών εξελοξής πιστοληπτικής ικανότητας είναι ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο από πολιτική άποψη. Το έχουμε παρατηρήσει και πρόσφατα κυρίως κατά τη διάρκεια συζητήσεων πολιτικών και εκλογικών. Ε, υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στην κοινή γνώμη. Εγώ θεωρώ ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι εκπροσωπούμε την Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη και τους Ευρωπαίους πολίτες, έχουμε ούτως ή άλλως το καθήκον να δώσουμε απαντήσεις. Οι οποίες θα είναι καινοτόμες, ισορροπημένες, λογικές, αλλά δεν πρέπει να Ρίψω κινδυνεύσουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι η συμβολή μας δεν αλλάζει το τρέχον πλαίσιο και ότι η τάση θα είναι να αφήσουμε τα πράγματα όσο έχουν σήμερα. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν καλό ουσιαστικά λόγω του σημαντικού πολιτικού θεσμικού ρόλου που διαδραματίζουμε εμείς εδώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολύ χρόνο για το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, αλλά ξέρω ότι θέλουν να ότι πρέπει να φύγουν κάποιοι συνάδελφοι για να ψηφίσουν σε άλλη επιτροπή. Η Ashley Fox, από ό,τι με ειδοποίησε, πρέπει να ψηφίσει σε μία άλλη ε, επιτροπή. Λοιπόν, ε, ο Ashley Fox, συγγνώμη, θα του δώσω λοιπόν το λόγο αν συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ντομινίτσι για τη δουλειά σας, για την ε, θέμα αυτό. Είπατε ότι το θέμα των οργανισμών επισκεπτικής ικανότητας έχει προκαλέσει ε, κάποια ε, εντύπωση, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να, κατηγορούμε τις ε, ε, του οργανισμού πιστολεπτική αξιολόγηση για το γεγονό ότι οι κυβερνήσει έχουν δαπανίσει υπερβολικά πάρα πολλά χρήματα, γιατί οι οργανισμοί αυτοί φαίνεται να έχουν, ε, οι οργανισμοί φαίνεται να έχουν εξουσία και να ελέγχουν τι κυβερνήσει. Αλλά γι' αυτό φταίνουν οι κυβερνήσει, γιατί έχουν δαπανίσει πάρα πολύ και έχουν ε, δανειστεί πάρα πολλά επί σειρά ετών. Και αυτό ισχύει και για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπω και για άλλε χώρε. Προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα να βγει από τις, ε, τα χάλια που έχει μπλέξει τα τελευταία 13 χρόνια. Δεν νομίζω λοιπόν, θα, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ε, αναλάβουμε τις ευθύνε μας ω πολιτικοί. Δεν φταίνε οι οργανισμοί επιστολεπτική αξιολόγηση που τώρα αγωνίζονται οι κυβερνήσει να ε, Τώρα σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέο, εγώ πιστεύω Είμαι κατά οποιαδήποτε μορφή ε, ε, unsolicited rating, ε, αξιολόγησης χωρίς να έχει ζητηθεί. Νομίζω ότι ο φόβος υποβιβασμού του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο στο να συμπεριφερθεί τόσο ε, αν θέλετε, διστακτικά και αυστηρά σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέο. Και το ίδιο ισχύει και οι άλλε κυβερνήσει. Και όλοι θα πρέπει να δανειζόμαστε λιγότερο. Δεν σύμφωνο με οποιοδήποτε είδου ευρωπαϊκό ίδρυμα που θα μπορεί να εκδίδει τέτοιε ε, αξιολογήσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες, γιατί είμαι βέβαιος ότι αν υπήρχε αυτό το Ίδρυμα, τώρα όλες οι χώρες θα είχαν τριπλό Α, γιατί θα υπήρχε πολιτική πίεση από τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα υπήρχε αξιοπιστία. Εκεί που συμφωνώ μαζί σας είναι ότι αν αν unsolicited rating θα πρέπει να δίδεται και να εκδίδετε όταν είναι κλειστές οι αγορές. Και γι' αυτό λοιπόν θα υποστήριζα μια σχετική πρόταση ότι οι αλλαγές σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση θα πρέπει να γίνονται μετά την, το κλείσιμο της αγοράς ε, της Παρασκευές ε, στην ε, Νέα Υόρκη. Νομίζω ότι είναι μια λογική και καλή πρόταση αυτή σε ό,τι αφορά τα θέματα αναλλαγής. Δεν υπάρχει υποστήριξη ούτε στο Συμβούλιο, ούτε στην Επιτροπή μας, κύριε Ντομινίτσι αν το σημειώσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει βέβαια συμφωνία να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να διαγραφούν όλες οι αναφορές στην εναλλαγή, γιατί είναι και ενάντια στις ε, δυνάμεις της αγοράς και είναι πολύ περίπλοκο και κανένα δεν βοηθάει στην τελική ανάλυση. Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι μια πρόταση και θα πρέπει να το συζητήσουμε και με το Συμβούλιο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Μπορεί Όταν χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, δύο οργανισμοί επιστολεπτικής αξιολόγησης, ε, ε, ο ένας να είναι μικρός. Ε, τώρα, αν θα χρησιμοποιηθεί το 10%, το 20%, όπως προτείνει ο κύριος Κλίντς, ή να το αφήσουμε στην ΕΣΜΑΝ, μια υποχρέωση αναφοράς για την κατάσταση ως προς τον ανταγωνισμό για να υπάρχει κάποια έτσι γνώση του που βρισκόμαστε Ξέρω ότι το Συμβούλιο ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την πρόταση αυτή και άρα ο συμβιβασμό θα είναι ε, εύκολος. Να σημειώσουμε όμως ε, ότι οι οργανισμοί πιστολεπτικής αξιολόγησης θα πρέπει να σημειώσουν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια ολιγοπόλια με δύο τέτοιου οργανισμούς. Θα πρέπει να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Τώρα, για θέματα αστικής ευθύνης. Δεν έχω πιστεί ότι υπάρχει οποιοδήποτε όφελος για να αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς και επίσης παραβιάζουμε τα καθεστώτα αστικής ευθύνης των 27 κρατών μελών. Ίσως λοιπόν αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι το κράτος μέλος έχει κάποιο καθεστώς για την αστική ευθύνη, αλλά εν πάση περιπτώσει να επαφίεται στα χέρια του κράτους μέλους, όπως έχει δηλαδή η κατάσταση στην παρούσα φάση. Δεν θυμάμαι, κύριε Ντομένιτσι, να αναφέρεστε, να αναφερθήκατε στο θέμα των αξιολογήσεων τρίτων χωρών. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέλθει στο καθεστώς της υποστήριξης που υποστηρίζει και ο κύριος Κλίντς. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια πιο μεγάλη περίοδο μεταβατική και θα πρέπει να προσέξουμε Προτού επιβάλλουμε ένα τέτοιο καθεστώς σε ε, δικαιοδοσίες άλλων κρατών, τρίτων κρατών. Θα υπάρχει αντίκτυπος και στο κεφάλι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες ήδη έχουν μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα κεφάλαια. Να μην δυσκολέψουμε περαιτέρω την ζωή τους. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο πρώτο και ευχαριστώ, λέει και δεν έχει έρθει ο εισηγητή του ΕΛΚ. Εκπροσωπεί κάποιο άλλο τον Ζων Πόλη, ίσω εσείς. Θέλετε να πάρετε το λόγο αργότερα, μάλιστα. Ο κύριο Κλίντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, συμφωνώ με τα εισαγωγικά σχόλια του κυρίου Ντομένιτζη και του Άσλι Φόξ ότι όντως πρόκειται για ένα πολιτικά πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και ότι θα πρέπει να προσέξουμε ακριβώς επειδή είναι τόσο πολιτικά ευαίσθητο το θέμα αυτό, να προσέξουμε λέγω να μην καταστούμε τελικά συναισθηματικοί σε ό,τι αφορά ε, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Να είμαστε ψύχρεμοι. Αυτό που είναι γεγονός, έχει δίκιο ο Άσλι, ότι τα κράτη-μέλη δεν περιήλθαν σε δύσκολες καταστάσει επειδή ε, ήταν κακές οι αξιολογήσεις τους. Όχι. Γεγονός όμως είναι ότι τα χρέη τα οποία ε, επιβαρύνουν τις χώρες προήλθαν και από τις ε, εν μέρη, εν τουλάχιστον, από τις λανθασμένες αξιολογήσεις. Άρα υπάρχει και μια εσωτερική συνάφεια η οποία όντως υφίσταται. Να εξετάσω τώρα τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν με τη σειρά με τη σειρά που τα ανέφερε και ο κύριος Ντομένιτσι. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το εθνικό, το δημόσιο χρέος. Δεν ε, πιστεύω ότι πρέπει να απαγορεύσουμε τα unsolicited ratings θεωρώ ότι το θέμα του δημόσιου χρέους ε, έχει να κάνει και με την υπερβολική εξάρτηση, το over-reliance. Αν μπορέσουμε να επιλύσουμε το θέμα του over-reliance, τότε αυτόματα θα λυθεί και το θέμα της αξιολόγησης ε, του δημόσιου χρέους. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι η απάντηση θα ήταν να δημιουργηθεί μια δημόσια αρχή ανεξάρτητη για την αξιολόγηση, γιατί αυτό είναι παράδοξο. Μια δημόσια τέτοια αρχή δεν πρόκειται να είναι ανεξάρτητη. Θα υπόκειται σε πολιτική πίεση. Συμφωνώ βέβαια με τον κύριο Ντομένιτσι ότι υπάρχουν θεσμικοί όροι, θεσμικοί, θεσμικά όργανα που μπορούν να αξιολογήσουν πάρα πολύ καλά την πιστοληπτική ικανότητα των χωρών. Όσα οι Εθνικές Τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μάλιστα αλλά θα ήταν λάθος να αναγκάσουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για παράδειγμα, να δράσει στον τομέα αυτό. Θα οδηγούσε σε διαφωνίες σχετικά με το αν θα ήταν σωστή ή όχι η αξιολόγηση της χύψη χώρας και αυτό θα έπλητε την ε, αξιοπιστία. Και δεν συμφωνώ να ιδρυθεί και ένα εθνικό ίδρυμα χρέους. Αυτό θα ήταν ένα πρώτο βήμα για τα ευρωμόλαγα. Αυτό με το μπλέκουμε με το θέμα των ε, οργανισμών αξιολόγησης πιστολεπτικής ικανότητα. Το δεύτερο θέμα που ανέφερε και ο κύριος Φόξ, το θέμα της εναλλαγή. Εγώ δεν είμαι υπέρμαχος τη εναλλαγή. Το πρόβλημα καταλαβαίνω ότι είναι η έλλειψη ανταγωνισμού. Μίλησα και και με διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων του DAX και κατάλαβα ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι οργανισμοί αυτοί θα ζητούν διπλάσια τέλη, διπλάσια, διπλάσια αμοιβή για τις ίδιες υπηρεσίες που α, χορηγούσαν ως τώρα. Αυτό καταδεικνύει τη μονοπωλιακή τους θέση και φυσικά δεν είναι θεμητό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον ε, η αρχή της εναλλαγής, ακόμα και αν τηρηθούν ε, οι προθεσμίες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, θα βοηθήσουν. Εγώ θεωρώ ότι όντως θα πρέπει να προδιαγράφεται σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται, πάνω από, δύο οργανισμοί να είναι ένας από τους δύο μικρός. Τρίτο σημείο. Σε ό,τι αφορά θέματα ευθύνης. Αντίθετα με τον Άσλι, και συμφωνώ απόλυτα με τον Ντομένιτσι, θεωρώ ότι θα πρέπει να εισαχθεί το σύστημα της αστικής ευθύνης, ωστόσο υπό τις αρχές ε, του κράτους δικαίου και όπως ήθιστε και στις υπόλοιπες ε, χώρες. Να μην υπάρξει βάρος, το αντιτροφή του βάρους απόδειξης. θα πρέπει να διαπιστώσουμε το εξή. Το θέμα δεν είναι να τιμωρηθούν ε, οι οργανισμοί επιστοληπτικής αξιολόγησης επειδή ε, εξέδωσαν μία αξιολόγηση που δεν μας άρεσε. Όχι. Τους ζητούμε όμως να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε περίπτωση που δεν θα τηρήσουν τις προδιαγραφές που ορίζονται με την νομοθετική αυτή διαδικασία. Και αν υπάρχει κάποια μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, της αξιολόγησης των διαρθρωμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Αν υπήρχε, είμαι βέβαιος, αυτή η ρύθμιση στο παρελθόν, θα είχαμε ε, κερδίσει κάτι. Για το μέλλον όμως θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι παραβιάσεις κατά του κανονισμού κατά της απαγόρευσης ε, σύγκρουσης συμφερόντων, θα είναι καταγγελτές, αλλά βάσει του υφιστάμενου του ισχύοντος ε, δικαίου, δικαίου που διαφέρει στα 27 κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει εναρμονισμένη νομική βάση. Τέταρτο σημείο σε ό,τι αφορά την υπερβολική εξάρτηση των οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Και εδώ ο συνάδελφος ε, ε, Ντομενίτσι αναφέρθηκε στην αναφορά της ΕΚΤ. Στο σημείο 4 να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η ίδια προδιαγράφει ότι οι οργανισμοί επιστολεπτικής αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και μάλιστα αναφέρει, τις, ε, αναφέρει τις οργανισμούς αυτούς ε, ονομαστικά. Αναφέρει βέβαια και άλλες πέρα από τις τρεις βασικές τέτοιες εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επενδυτές, ιδιαίτερα οι, θεσμικές, οι θεσμικοί επενδυτές, αναλαμβάνουν την ευθύνη τους και δεν θα πρέπει να σας απαλλάξουμε από την υποχρέωση την οποία, στην οποία υπόκεινται για το σε ποιες αξιολογήσεις βασίζονται. Τώρα κατά πόσον ε, θα ένα χρονικό περιθώριο 6 μηνών, 3 χρόνια, ε, Γκοζές ντομενιτς εγώ το αφήνω ανοιχτό, δεν νομίζω ότι είναι το καθοριστικό πέμπτο σημείο τώρα. Ε, θέματα μεθοδολογίας. Έγινε διευκρίνηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα δεν είναι το περιεχόμενο, η ουσία να ελέγχεται από την ΕΣΜΑ. Όχι, η διαδικασία θα πρέπει να ελέγχεται και αν οι μέθοδοι τροποποιούνται, θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να κοινοποιούνται στην ΕΣΜΑ και η ΕΣΜΑ έχει χρόνο ένα μήνα για να αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει, αν θεωρείται εγκεκριμένη τροποποίηση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια καλή λύση. Τώρα, συγκεκριμένα... Θα πρέπει να προσέξουμε προκειμένου το επιχειρηματικό μοντέλο που έχει επιλέξει η... ο Οργανισμός Προληπτικής Αξιολόγησης ε, ε, δυσκολεύεται, δυσχεραίνεται. Τελευταίο σημείο, το θέμα Τη σύγκρουση συμφερόντων και κυρίως τη συμμετοχή στις, ε, στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοτικής ικανότητας. Ε, ακούσαμε πολλά και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη συμμετοχή. Το πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως προκύπτει είναι αν υπάρχει συμμετοχή σε ταμεία δικτών, μπορεί να ξεπεραστεί το 5%. Και τελευταίο σημείο που ήθελα να αναφέρω, το ανέφερε και ο Άσλι Φόξ. Λυπάμαι ιδιαίτερα που η ρύθμιση για τις τρίτες χώρες τα τελευταία 1,5-2 χρόνια έχει τροποποιηθεί γιατί υπήρχε μια τέτοια ε, ρύθμιση, ένα endorsement, αλλά η ερμηνεία αυτού που υπήρχε τότε έχει αλλάξει πλέον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Δυστυχώς, γιατί αν ε, ε, επιμείνουμε αποκλειστικά σε θέματα εξίσωσης, υπάρχει ο κίνδυνος Ακόμα και οι οργανισμοί που είναι καταχωρισμένοι και εγκεκριμένοι στην Ευρώπη θα κληθούν να επιβεβαιώσουν αξιολογήσεις εκτός της Ευρώπης. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στέγνωμα των αγορών, μπορεί να οδηγήσει την Ευρώπη Μπορεί να, αν θέλετε, αν είμαστε αισιόδοξοι, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προστατεύσει την Ευρώπη. Αφετέρου, μπορεί και να την απομόνωνε, σαν ένα κάστρο, αν θέλετε. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί από την αρχή το επιβεβαιώνω αυτό. Ε, άφησε να συμμετάσχουν και οι σκιώδεις ε, και αυτό οδήγησε σε πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Ε, thank you. ευχαριστώ. Φιλίπ, ευχαριστώ. Όπως είπες, Σάρον, αντικαθιστώ τον Πασκάλ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον Βόλφ. Αυτά που είπε στον εισηγητή, να τον ευχαριστήσω, διότι συνεργάστηκε και με τους Κιώδης και έτσι έγινε πολύ καλή δουλειά. Ο Άσλεϊ άρχισε με κάποια πολιτικής φύσεως σχόλια. Και εγώ το ίδιο θα κάνω. Βαρέθηκα να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όλο τα ίδια και τα ίδια λέμε. Η κρίση είναι κάτι το οποίο οφείλεται στους οίκους αξιολόγησης, αλλά είναι όχι, για, καλή, για κακή, κακοδιαχείριση των κυβερνήσεων. Εύκολο είναι να υιοθετήσουμε ή το ένα ή το άλλο επιχείρημα. Είπε λοιπόν ο Άσλεϊ, θα πρέπει να έχουμε αυτούς τους οίκους ώστε να κάνουν δουλειά τη δουλειά τους οι κυβερνήσεις. Το αντίθετο, πώς θα το επιτύχουμε. Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιονότησης αποτελούνται από άτομα τα οποία ε, δεν είναι υπεράνθρωποι, ενώ στις κυβερνήσεις συμμετέχουν ε, ανθρώπινα όντα που λανθάνουν πολλές φορές. Τι κάνουμε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι να κάνουν τη δουλειά τους σωστά οι κυβερνήσεις και να μην ασχολούμεθα υπερμέτρως με αυτές τους οίκους. Εν πάση περιπτώσει, όντως είχαμε τέτοια προβλήματα διαχείρισε κάποιες χώρες αλλά και αυτοί οι οίκοι με τα σχόλια που έκαναν και που ήταν λαθασμένα πολλέ φορέ οδήγησαν σε λαθασμένε συμπεριφορέ. Και μετά λένε Απαπα, συγγνώμη. Εν πάση περιπτώσει, ουδή αναμάρτητο, ούτε η μεν, ούτε η δε. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Δεύτερον, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι να έχουμε μια δημόσια τέτοιο ε, ε, οργανισμό, ένα ίδρυμα και την υπερεξάρτηση. Αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Εάν κατορθώσουμε να μην έχουν σχεδόν αυτόν τον επίσημο ρόλο αυτή η οίκη αξιολόγησης που έχουν την εντύπωση ότι παρέχουν ένα κοινό αγαθό, εάν μπορέσουμε να τις κάνουμε να υιοθετήσουν το ρόλο τους έτσι όπως πρέπει να είναι, πιστεύω ότι η εναλλακτική λύση του Ιδρύματος ή της δημόσιας αυτού ε, οργανισμού θα πρέπει να παραμείνει. Εάν δεν θέλουμε να τους δώσουμε αυτό το ρόλο, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της αξιολόγησής τους θα είναι λιγότερες και εδώ χαιρετίζω τις προτάσεις του Άσλεϊ και του Βόλφο όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Εάν λοιπόν μειώσουμε τον επίσημο ρόλο τους και έχουμε και εισαγάγουμε το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας, θα έχουμε καλύτερη ισορροπία. Uh, uh, Επίσης, κάτι αναφέρθηκε από τον Διόγκο Φέο για Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον δανεισμό. Εγώ δεν συμφωνώ. Πρόκειται για την εφαρμογή όντως των ευρωομολόγων. Αν το θέλουμε και αν θέλουμε να κάνει κάτι τέτοιο η Ευρώπη, δεν νομίζω ότι θα πρέπει εδώ το θέμα αυτό να το συζητήσουμε από κοινού με τους οίκους αξιολόγησης. Κάποια άλλα σημεία που θεωρούμε σημαντικά, σύντομα θα αναφέρω. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ίσως περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμούς. Το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι μηχανικός αλλά κάτι το οποίο να καταλαβαίνει ο κόσμος παρά αυτές τις επιστολές που έχουν χιλιάδες συμβολισμούς και δεν καταλαβαίνει. Τώρα αφορά τη μεθοδολογία. Το ανέφερε ο εισηγητής, θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη όλους τους κινδύνες και να αρχίσουμε να λαμβάνουμε υπόψη τους κινδύνες που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν από η υπερτίμηση ή από η κακή εκτίμηση ή υποτίμηση και ακόμη για θέματα ευρωστίας των επιχειρήσεων. Πέρσι είχαμε πλημμύρες πολύ στην Ταϊλάνδη. Και σταμάτησαν κάποιες επιχειρήσεις να εργάζονται κυρίως στα θέματα της ηλεκτρονικής, είχαμε κάποια προβλήματα. Θα πρέπει τέτοιου είδους ε, Επιχειρήσει που μας ενημερώνουν για τους κινδύνους που μπορούν να υπάρξουν και επηρεάζουν την οικονομία, του λαμβάνουμε υπόψη. Στο άρθρο 8 γίνεται λόγος για κάποιες οικονομικές ε, απαιτήσει, οικονομικά μέτρα. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή επιτροπή επενδυτών και καταναλωτών και αυτό είναι το όλο θέμα. Ποιο πληρώνει αυτέ του οίκου αξιολόγηση. Νομίζω ότι εδώ σε συνδυασμό με ανταγωνιστικότητα και λιγότερο σημαντικό και επίσημο ρόλο για αυτές και αν χειριστούμε το θέμα των οικονομικών αυτών των επιχειρήσεων θα έχουμε ε, περισσότερη ε, ειλικρίνεια στο επίπεδο τους και αυτό το χρειαζόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να μελετήσει ε, όλα τα κονδύλια τα οποία δίδονται και τα μοντέλα βάσει τα οποία δίδονται η Κομισιόν. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε είναι να εμπλακούν και στην πολιτική αυτή η ε, οίκη αξιολόγησης. Αυτό δεν το υποστηρίζουμε. Ο καθένα θα πρέπει να μείνει στα πλαίσια του ρόλου του. Αν θέλουν να γίνουν πολιτικοί, ας ε, είναι υποψήφιοι στι επόμενε εκλογέ. Τώρα, η υπερβολική εξάρτηση και η εναλλαγή. Η πρόταση επιτροπή είναι κάπως επαρκής, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε ένα πιο εύκολο σύστημα και καθεστώ εναλλαγής να προτείνουμε βάσει τροπολογιών τις οποίες θα καταθέσουμε. Αλλά και υπάρχουν ακόμη θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε, πράγμα το οποίο και πάλι πρέπει να πω ότι δεν είναι ε, ασύμβατο με τα θέματα της αντιγωνιστικότητας. Προς το παρόν σταματώ εδώ και ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ. Ήρθε ο Ζων Πολ και του δίνω αμέσω το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Έφτασα τελευταίο. Ζητώ συγγνώμη διότι είχα δύο άλλε ανηλυμένε υποχρεώσει. Συνάντηση με τον πρόεδρο Βον Ρομπάι και βεβαίω δεν μπορώ εγώ να επηρεάσω τώρα την ώρα του ραντεβού. Ήδη με τον εισηγητή δήμερος, Είχαμε αναφερθεί σε κάποια από αυτά τα θέματα. Δεν θα τα επαναλάβω. Το πρώτο θέμα το οποίο μας ε, απασχολεί είναι κοινό θέμα. Να μην υπάρχει υπερβολική εξάρτηση όσον αφορά τους βαθμούς που δίδουν κατά την αξιολόγησή τους αυτή η Δεύτερο θέμα, μηχανισμός αναλλαγής. Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος διότι νομίζω ότι δεν θα καταλήξουμε σε κανένα θετικό και προσδοκόμενο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί ολιγοπόλιο ή ιδιοπόλιο υπέρ των δύο μεγάλων ε, τέτοιων οίκων. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Ξέρω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα προσφυλές στον Επίτροπο και εγώ δεν θέλω να στενοχωρώ το φίλο μου το Μισελ Μπαρνιέ, εν πάση περιπτώσει δεν συμμερίζομαι για το θέμα αυτό τη Επιτροπή. Υπάρχει επίση το θέμα τη αστική ευθύνη νομίζω θα πρέπει να κάνουν διαφοροποίηση μεταξύ της ευθύνη της αστικής και της ε, ευθύνη της πειθαρχικής για πειθαρχία. Όταν δεν σέβεται τους κανονισμούς ο οίκος υπάρχουν και προβλέπονται κυρώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να υπάρχει και επίπτωση στην αστική ευθύνη εάν δεν συντρέχουν οι λόγοι. Πιστεύω λοιπόν ότι οι κανόνες που θα εφαρμόζονται θα πρέπει να, είναι αυτοί που ισχύουν στις διάφορε χώρε και για την Γαλλία για να μπορέσει κανείς ε, ε, να κατηγορήσει κάποιον ή να του προσδώσει μάλλον αστική ευθύνη θα πρέπει να έχει σύμφωνα με τον νόμο τώρα όσον αφορά την αντιστροφή του βάρους απόδειξης και εδώ θα πρέπει να είμαστε μετριοπαθείς διότι εάν υπάρξει πλήρης αντιστροφή του βάρους απόδειξης θα έχουμε πολλαπλές διαφορές που θα κάνουν τους πάντες να χάσουν χρόνο για ένα πολύ μέτριο ε, αποτέλεσμα. Και οι θα πούνε συνέβη αυτό που συνέβη, είναι λάθος του οίκου αξιολόγησης. Εάν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να θέσει ένα αμφιβόλο την αξιοπιστία του οίκου αυτού, θα πρέπει να πει κατά πρώτο λόγο κατά την άποψή του που έσφαλε ε, ο οίκος αξιολόγησης, πώς το διασυνδέει με το πλήγμα το οποίο υπέστη και να ακολουθήσει τη δικασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ούτε και εδώ θα πρέπει να είναι υπερβολικά εύκολος ο τρόπος τον οποίο να μπορεί κανείς ε, να ζητάει την οποδήποτε διόρθωση. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ποσά τα οποία επενδύθηκαν, ποια είναι η ζημία που υπέστη ο και κτλ, κτλ. Αν υπάρχει ρευστότητα, αν υπάρχει κτλ. Τώρα, όσον αφορά τις τρίτες χώρες. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξανανοίξουμε τη συζήτηση η οποία ολοκληρώθηκε για αυτό το θέμα στα δύο πρώτα κείμενα. Δύο λόγια θα πω μόνο. Από πολιτικής πλευράς όσον αφορά την αξιολόγηση του δημοσίου χρέους. Πολλοί προτείνουμε οι οίκοι αυτοί να μπορούν να αξιολογούν τις χώρες, αλλά να δίδουν την απόφαση, να κάνουν την αξιολόγησή τους σε ημερομηνίες βάσει χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα είναι γνωστό στις κυβερνήσεις, ώστε να μην δίδονται αυτές οι αξιολογήσεις στην παραμονή της ψήφισης του προπολογισμού ή την παραμονή ενός ε, Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Είδαμε τι συνέβη την Πορτογαλία. Για την ε, αξιολόγηση λοιπόν ε, και την βαθμολόγηση των οίκων αυτών να διατηρηθεί, αλλά ας πούμε φέρει την πρώτη Παρασκευή κάθε αρχής ενός τριμήνου, μετά το κλείσιμο των αγορών, την Παρασκευή το απόγευμα, εν πάση περιπτώσει κάποια συμφωνία να βρούμε με τρόπο ώστε αυτή η οίκη αξιολόγησης ίσως και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που αφορώνται από αυτήν την αξιολόγηση να μπορούν να αιτιολογήσουν μία κατάσταση και να πούνε και ποια είναι η δική τους αξιολόγηση. Αυτά είναι τα σημεία που ήθελα να αναφέρω. Η συνεργασία μας με τον εισηγητή ήταν εξαιρετική και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα κείμενο ποιότητος το οποίο θα συμπληρώσει τα δύο πρώτα κείμενα τα οποία εμένα με ενδιαφέρουν και θέλω να εφαρμοστούν κατά γράμμα από την ΕΚΑ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Άλλοι ομιλητές. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία του. Νομίζω ότι πραγματικά τις τελευταίες εβδομάδες ε, φρόντισε πάρα πολύ τους ε, εισηγητές, τους και εισηγητές σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μαζί τους. Θα ήθελα εξ αρχής να προσθέσω ότι σε κάποια ε, ζητήματα υποστηρίζει τον συνάδελφο Φέγιο, ο οποίος έχει φύγει ήδη για Πορτογαλία για τα θέματα ε, εναλλαγής, ε, για θέματα ε, ανταγωνισμού. Θα καταλάβετε όμως ότι δεν συμφωνώ σε ό,τι αφορά ε, την, σύμφωνα με τον κύριο Φέγιο ό,τι αφορά τα θέματα των, ε, του Ιδρύματος ε, για τα χρέη. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία σε ό,τι αφορά τους οίκους αξιολόγησης, ε, μείωση της συγκέντρωσης της αγοράς, αποφυγή και μέτρα κατά της ε, σύγκρουσης συμφερόντων και ε, μέτρα κατά της τυφλής εμπιστοσύνης. Και, θα, και πρέπει να σκεφτούμε και πάλι το θέμα του δημόσιου χρέους σε ό,τι αφορά θέματα αστικής ευθύνης ε, των οίκων αξιολόγηση. θεωρώ ότι είναι πολύ σωστό βήμα. Σε ό,τι αφορά τη διευκρίνηση για την ευθύνη δυναστική, θεωρώ ότι χρειάζεται μια τέτοια πρόβλεψη επιγόντως, αλλά θα πρέπει να γίνει μια περαιτέρω διευκρίνηση και να διασφαλίσουμε ότι ε, το τεκμήριο αθωότητας το οποίο ισχύει γενικά στο νομικό μας σύστημα ισχύει και για τις οίκους αξιολόγησης. Ε, επίσης, σε ό,τι αφορά τους αυτοματισμούς ε, για τα, τους οίκους αξιολόγησης θεωρώ ότι θα πρέπει να μειωθούν για να μειωθεί και η υπερβολική εξάρτηση στους οίκους αξιολόγησης, από τους οίκους αξιολόγησης. Ο ανταγωνισμός είναι αυτό που λείπει κατεπηγόντως σήμερα από την αγορά, αλλά ως ρυθμιστική αρχή δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε να υπάρχει ανταγωνισμός ε, γιατί τελικά μόνο μία έκθεση αξιολογικού οικοαξιολόγησης ε, ε, θα ε, επικρατήσει. Αλλά αν κανείς δεν μπορέσει να, να έχει εμπιστοσύνη στους νέους αυτούς ε, θεσμούς αξιολόγηση, αξιολόγησης, δεν θα έχει νόημα δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός. Ε, τώρα, κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν ιδρύματα. Αν ε, αποφασίσουμε να λάβουμε μέτρα για τον ανταγωνισμό μεταξύ των ε, οίκων αξιολόγησης που υφίστανται, θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα τα μέτρα αυτά. Ο περιορισμός της, του μεριδίου στην αγορά δεν είναι εφαρμόσιμος, θεωρώ. Θα πρέπει σίγουρα να αποφεύγουμε σύγκρουση συμφερόντων, αλλά θεωρώ ότι το σχέδιο έκθεσης εδώ δεν πάει αρκετά μακριά. Αν αγοράσω αύριο μία μόνο μετοχή, μεταξύ της μιας επιχείρησης και ενός οίκου αξιολόγησης, ε, τι θα ισχύει τελικά. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και αυτή η πρόβλεψη, αυτός ο κανονισμός θεωρώ ότι γίνεται ακόμα πιο αμφισβητήσιμος όταν ε, εισαχθεί η αρχή της αναλογής. Αν υπήρχε ε, σήμερα μια πληθώρα εικοναξιολόγησης για όλα, τονίζω όλα τα προϊόντα, θεωρώ ότι η αναλλαγή θα ήταν ένα καλό ε, μέτρο, αλλά πω έχει η κατάσταση σήμερα. Δεν θεωρώ ότι είναι εφαρμόσιμα τα μέτρα αυτά και σε ό,τι αφορά αυτή την ε, περίοδο cooling off. Αν οι τρία, αν τρι, τρεις μεγάλοι οίκοι ε, αξιολόγηση έχουν μπλοκαριστεί ε, λόγω της περίοδου cooling off. Τι θα γίνει με τους μικρούς οργανισμούς. Και επιπλέον, σε θέματα εναλλαγής μπορεί να υπάρχουν και άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Αστάθεια των αγορών, αυξημένη μείωση της ποιότητας των εκθέσεων αξιολόγησης. Θεωρώ λοιπόν συνοπτικά ότι σε ορισμένα σημεία θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη να γίνει μεγαλύτερη συζήτηση και ελπίζω οι τροπολογίες μου να εισακουστούν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον πίθεσή μου. Ja, lieber Burkhard, das ist jetzt seit langem das erste Mal. Είναι η πρώτη φορά που διαφωνώ μαζί σου, συνάδελφε. Και να σου εξηγήσω και γιατί. Γιατί Αυτό που είναι αυτονόητο για κάθε υπάλληλο τη φαρμακοβιομηχανίας, ότι δεν μπορεί να έχει, για παράδειγμα, ε, μετοχές τη ε, ε, επιχειρήση αυτή, ακόμα και αν δεν εργάζονται άμεσα με το προϊόν αυτό, το οποίο περνάει από αξιολόγηση, αναγκάζονται από τις επιχειρήσεις αυτές είτε να πουλήσουν τις ε, μετοχές τους ή να μην τις αγοράσουν. Και γιατί, γιατί, σε ένα, γιατί να ισχύει κάτι διαφορετικό εδώ πέρα, που είναι πολύ πιο μεγάλο το οικοδόμημα. Γιατί να ισχύει κάτι διαφορετικό από για τους υπόλοιπους υπαλλήλου να προσέξουμε μια επιχείρηση που κάνει τέτοια αξιολόγηση, να μην βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση τέτοια, σε μια τόσο ευάλωτη κατάσταση, να μην έχει και υπαλλήλου που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση σύγκρουση συμφερόντων. Για να αποφευτούν λοιπόν οι συγκρούσει συμφερόντων, θα πρέπει τα μέλη και οι υπάλληλοι των οίκων αξιολόγηση, όχι μόνο όπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να μην έχουν έμεσα ή άμεσα συμφέροντα στην επιχείρηση, αλλά να μην έχουν και διαθρωμένα χρηματοπιστωτικά μέσα σε ό,τι αφορά την επιχείρηση αυτή. Και αυτό που δεν έλαβε υπόψη δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παράλληλη σύγκρουση συμφερόντων σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση εθνικών ομολόγων. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ανάλογα θα πρέπει να επεκταθεί αυτή η ρύθμιση και σε ό,τι αφορά τα εθνικά ομόλογα. Όλα τα μέλη και οι υπάλληλοι των οίκων αξιολόγηση δεν θα πρέπει να έχουν ούτε συμφέροντα σε εθνική ομόλογα, ούτε σε διαθρωμένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Στο σημείο λοιπόν αυτό οι απόψει μα είναι διαμετρικά αντίθετε. Και τέλο ναι, είναι ενδιαφέρον. Τέλο, θα ήθελα να επισέλθω και σε ένα άλλο σημείο, το οποίο ίσω να έκανε λιγότερη εντύπωση, αλλά μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Δεν το ακούσαμε ιδιαίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και αξιολόγηση στο website τους να δημοσιεύουν πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις και για τα μέσα χρέους που έχουν ζητήσει ε, διεξαγωγή και κατάρτιση εκθέσεων. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά να έχουμε υπόψη μας και το συμφέρον εκείνου που θέλει να δώσει μια τέτοια εντολή. Η δημοσίευση προτού εκδοθεί, δημοσιευτεί αυτή η έκθεση, θα τον εκθέσει σε κερδοσκοπία της αγοράς. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εποπτική αρχή, να ενισχύσουμε την ΕΣΜΑ, πολύ ωραία στο σημείο αυτό, να υπάρχει υποχρέωση αναφοράς για μια τέτοια αξιολόγηση, για μια τέτοια επιχείρηση που θέλει να εκδώσει τέτοια έκθεση, αλλά να μην ε, δημοσιεύεται υποχρεωτικά εκ των προτέρων αυτή η πρόθεση έκδοσης έκθεσης. Νομίζω μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ελέγχου, αλλά από την άλλη να λάβουμε υπόψη για τα συμφέροντα του πελάτη που ζητάει έκδοση. Και τελείωσα, κυρία Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ και ποιος θέλω, θέλει να μιλήσει. Ουντώ. Ja, vielen Dank, äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θυμάμαι το πνεύμα στο οποίο συζητήθηκαν στην τελευταία θητεία ε, η οίκη αξιολόγηση. Ε, ο συνάδελφος Γκοζές είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ο συνάδελφος Κλίντς. Και με ενοχλεί το εξή και σας το λέω ε, ανοιχτά ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε ε, με τους οίκους αξιολόγησης είναι μάλλον κυκλικός. Εμείς ως σοσιαλδημοκράτες τότε για τις εκθέσεις αυτές ε, στην προηγούμενη θητεία προσπαθήσαμε να δώσουμε ε, μία σαφή διάσταση να υπάρξει μία καλύτερη ρύθμιση και να ανοίξει η πόρτα για μία εναλλακτική λύση, για μία ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση ενδεχομένω. Τότε οι συνάδελφοι δεν ήταν δεθμένοι να προχωρήσουν. Γι' αυτό λοιπόν ήταν πολύ προσεκτική διατύπωση με μία αντολή ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο μεταξύ έχουμε περάσει την ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Το θέμα λοιπόν έχει αλλάξει και στο Συμβούλιο στις Πρωτεύουσες και εδώ στην Επιτροπή. Όλοι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε παραπέρα και να πούμε ότι όχι, θα πρέπει να υπάρχει σαφής ρύθμιση, αξιοπιστία, διαφάνεια αστική ευθύνη, ποιο είναι υπεύθυνο γιατί και θέλουμε να δημιουργηθεί και μια εναλλακτική για να σταματηθεί αυτή η μονοπωλιακή κατάσταση. Ακούγοντα λοιπόν τι γίνεται σήμερα, θεωρώ ότι και πάλι αρχίζουμε θεματικά να ξαναπέφτουμε, κατηφορίζουμε. Είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί στην ε, επιχειρηματολογία και αυτό μου έκανε εντύπωση στο θέμα του ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Από πού προερχόμαστε όμως, από μια κατάσταση όπου έως τώρα το προϊόν της αξιολόγησης θεωρείται ε, μία απλή έκφραση άποψης κατά το αμερικανικό μοντέλο και κανείς ε, δεν ευθύνεται για τίποτα γιατί ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης τους και η όλη διαδικασία νομικά δεν θεωρείται ως παροχή υπηρεσίας. Δεν υπάρχει ε, σύμβαση ευθύνης. Από αυτή την κατάσταση προερχόμαστε και ακούγοντας τη σημερινή συζήτηση έχω την εντύπωση ότι κινούμαστε σε ένα περιβάλλον, σε μια ατμόσφαιρα όπου θέλουμε να αποφύγουμε μια ρύθμιση. Και ε, η αρνητική γνώμη για μια ευρωπαϊκή θεσμική αρχή. Ακούω για, από τη Φραγκφούρτη ότι υπάρχει υπάρχουν προβλήματα, θεωρώ ότι αυτή η απόρριψη της πρότασης αυτής είναι πολύ πρόημη. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε εναλλακτικέ και νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσουμε και να υποστηρίξουμε τον εισηγητή που προσπαθεί να καταρτήσει μια τολμηρή έκθεση. Αυτό απευθύνω ως έκκληση προς τους συναδέλφους. Okay, anybody Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Καταστρέφω τα πάντα εδώ πάνω στην έδρα. Στο μεταξύ θα ήθελα να πω μερικά πράγματα κι εγώ ίδια. Έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες σε διάφορα σημεία για να επισημάνω αυτά που θεωρώ σημαντικά. Όσον αφορά το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ανεξαρτησία, όπως το ανέφεραν και άλλοι. Όσον αφορά το ζήτημα των εθνικών χρεών, των δημοσίων χρεών, δεν πρέπει να υπάρχει πολιτική πίεση ή οτιδήποτε που θα σήμαινε ότι η αξιολόγηση που δίδεται δεν είναι σωστή και ότι δεν ε, λαμβάνει υπόψη όλους τους ε, σωστούς παράγοντες. Καλό είναι να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα επίσης για την ε, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ώστε να μην ακούμε επικρίσεις του κατά πόσο γίνονται σε πολιτικά σημαντικές στιγμές και κατά πόσο έχουν κάποια βάση κάποιες θεωρίες συνωμοσίες ε, το να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα και να κατανοούν όλοι πότε βγαίνουν οι αξιολογήσεις όταν κλείνουν οι αγορές πιστεύω ότι αυτό έχει νόημα Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι οι εταιρείε δεν θέλουν επιπλέον κόστη και ότι σε όλες τις αγορές θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνέχεια όσον αφορά τον τρόπο δημοσιοποίηση των αξιολογήσεων και παραγωγή των αξιολογήσεων, να μην έχουμε αλλαγή των αξιολογήσεων επειδή άλλαξε ο οίκο αξιολόγηση. Έχω κάποιε αμφιβολίε όσον αφορά την αναλλαγή. Έχω υποβάλει τροπολογίε για την αναλλαγή ω την λιγότερο κακή επιλογή. Αυτό ο κύκλο αναλλαγή που προτείνεται από την Κομισιόν κοιτώντα ε, τι στιγμέ. Ε, ε, όπου πρέπει να γίνονται εξολογήσεις, δεν φαίνεται να μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά. Ε, αν είχα την επιλογή θα επέλεγα καμία εναλλαγή. Αυτό προσφέρω εγώ ως τη λιγότερο κακή επιλογή. Εγώ λοιπόν θα υποστηρίξω τη γραμμή που της ομάδας Alde και του Wolf Clint. Ε, αν κοιτάξουμε αυτό το να προσπαθούμε να ξεφορτωθούμε την υπέρμετρη εμπιστοσύνη, ε, αυτό πρέπει να το δούμε σε όλους τους τομείς. Δεν μπορούμε να το επιλύσουμε πλήρως με ένα κανονισμό, μάλλον καθόλου με τα όσα επιβάλλουμε στους οίκους επιστοληπτικής αξιολόγησης. Θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε με το CRD, με στο MIFID. Προσπαθούμε να τα πράξουμε όλα αυτά δεν είναι προφανές για όλους. Για παράδειγμα στο CRD όπου προτείνουμε να συμπεριλάβουμε ε, ασκήσεις benchmarking ε, ε, ώστε να συγκρίνουμε τραπεζικά μοντέλα και άλλα πράγματα. Έτσι προσδίδεται μεγαλύτερη διαφάνεια, άλλα πράγματα δηλαδή, τα οποία μπορούν να αρχίσουν να λαμβάνουν υπόψη επενδυτές εκτός από τις επιστολήπτικες αξιολογήσεις. Κοιτώντα το σκιώδε τραπεζικό σύστημα και την πολυπλοκότητα των τίτλων και κατά πόσο θα υπάρξει ή όχι παρέμβαση όπως συζητήσαμε χθε στο πλαίσιο του MIFID και όλα αυτά θα αποτελέσουν πρόληψη της υπερβολικής εμπιστοσύνη τη αξιολογή, γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση, μεγαλύτερη τυποποίηση σε ορισμένου τομεί, μεγαλύτερη διαφάνεια όχι μόνο στον τρόπο λειτουργία των οίκων ελληνική αξιολόγηση, αλλά και στη γενικότερη νομοθεσία. Αλλά δεν μπορούμε να καταργήσουμε την εμπιστοσύνη στις αξιολογήσεις εάν δεν προχωρήσουμε περισσότερο στην οδό που έχουμε ήδη ξεκινήσει και με άλλες νομοθεσίες ίσως να έχουμε δύο παράλληλες οδούς ε, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα λειτουργήσει μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ο διάλογος που άκουσα όσον αφορά την απαγόρευση της, ε, ε, του να έχει κάποιος μετοχές. Πρέπει να φροντίσουμε να το ορίσουμε σωστά. Θα έχουμε δείκτες και CDS και hedge funds και ίσως να είναι εύκολο κατά λάθο κάποιος να είναι δικαιούχος ενός τίτλου σε ένα σύνολο με το, μετοχικού κεφαλαίου διότι μπορεί να είναι έμεσα τα συμφέροντα. Εάν πρόκειται να ακολουθήσουμε τέτοια οδό θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι σαφές ότι αν το holding υπάρχει ως κάτι τυχαίο, ως περιστασιακό index, hedge ή κάτι τέτοιο, ότι δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, διότι δεδομένως της πολυπλοκότητας των προϊόντων που υπάρχουν, θα ήταν πολύ δύσκολο να καταργήσουμε όλα αυτά. Αυτά είχα να πω. Δίνω λοιπόν το λόγο ξανά στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ομιλίες τους. Πολύ, χρήσιμες, ε, πολύ χρήσιμα τα σχόλια και συνεισφέρουν σημαντικά στη συζήτηση. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το σημείο στο οποίο είχα φτάσει ολοκληρώνοντας την εισαγωγή μου. Ξεκινώ από την αναφορά σε μια αξιολόγηση του, των ειδησιών των κανονισμών. Ενδέχεται να έχει δίκιο ο συνάδελφος Γκοζές όταν υποστηρίζει ότι ίσως εάν είχε εφαρμοστεί αποτελεσματικά το κανονιστικό πλαίσιο που ήδη υπάρχει, ενδεχομένως δεν θα χρειαζόμασταν αυτόν τον νέο κανονισμό. Η δική μου απόψη είναι λίγο διαφορετική, ωστόσο σέβομαι τη δική του. Θεωρώ ότι η εφαρμογή του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου αποτελεί σημαντική πτυχή. Ωστόσο, το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτός ο νέος κανονισμός μπροστά μας και τον συζητάμε. Αυτό συμβαίνει διότι έχουν γίνει και συνεχίζονται διάφορες συζητήσεις ε, παρατηρείται ευαισθητοποίηση σε κάποιο επίπεδο και μας έχει προειδοποιήσει η Κομισιόν αλλά μας είχε προειδοποιήσει ήδη και ο συνάδελφος Κλίντς με την ε, ίδια πρωτοβουλία έκθεσή του να δώσουμε νέες προτάσεις. Έχετε δίκιο. Πρέπει να προσέξουμε, κύριε Μπούλμαν διότι αν υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση και αυτή η απέτηση να δώσουμε νέες απαντήσεις, αλλά ταυτόχρονα αυτές οι απαντήσεις που εμείς δίνουμε γίνονται αντιληπτές ε, από την κοινή γνώμη ως μη επαρκής, εμείς ως κοινοβούλιο και εμείς ως πολιτικές δυνάμεις, πολιτικοί εκπρόσωποι σε αυτό το κοινοβούλιο, εμείς θα πληρώσουμε το τίμημα. Και εμείς θα ακούσουμε τις επικρίσεις. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι μου είναι να συνεχίσουμε τις εργασίες μας ώστε να προσπαθήσουμε να δώσουμε αποτελεσματικές απαντήσεις αλλά και απαντήσεις τολμηρές σε σχέση με τα προβλήματα που έχουμε ενωπιών μας. Εγώ θεωρώ ότι η αρχή που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία είναι μια φιλελεύθερη αρχή είναι η ανάγκη ύπαρξης πολυφωνίας και πολλών διαφορετικών απόψεων που θα είναι δυνατόν να συγκρίνουμε, να αντιπαραβάλουμε ώστε να καταλήξουμε στις πιο σωστές αξιολογήσεις και στις πιο εξισορροπημένες αξιολογήσεις. Αυτό αφορά τόσο τις αγορές γενικότερα όσο και το ειδικότερο πιο συγκεκριμένο πρόβλημα που συζητήθηκε ιδιαίτερα πολύ σήμερα το πρωί της αξιολόγησης των δημοσίων χρεών. Εγώ συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι δεν πρέπει και δεν μπορούμε να, δώσουμε, να δίνουμε την εντύπωση ότι ε, παραβλέπουμε την ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά τη συσσόρευση υπερβολικού χρέους, αλλά δεν συζητάμε αυτό. Και δεν είναι αυτή η άποψή μου. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν εμείς ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο θέλουμε να αναλάβουμε ένα καθήκον και μια ευθύνη και όσον αφορά την εκπόνηση εναλλακτικών μεθόδων και τη διατύπωση επικρίσεων και αξιολογήσεων όσον αφορά την αξιοπιστία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Εάν όμως δεν το πράξουμε, και εγώ θα σας το πω με απόλυτη ειλικρίνεια και πολύ καθαρά, υποψιάζομαι ότι κατά κάποιο τρόπο μας βολεύει. Ότι δηλαδή δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και αφήνουμε τους οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης να έχουν την όλη ευθύνη την αναλαμβάνουν ευχαρίστως οι οίκοι πιστοληπτικής σε αυτή την ευθύνη. Α μην υπεκτιμάμε το πώ του δίνεται δωρεάν τόσο πολύ δύναμη επί των δημοσίων χρεών σε συγκεκριμένε στιγμέ, χωρί να λαμβάνουν υπόψη τι προκυκλικέ επιπτώσει. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αναλαμβάνουμε κάποιες ευθύνες διότι μας κουράζει να μελετήσουμε εναλλακτικέ μεθόδους. Αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν είναι ικανό κριτήριο για να μην το πράξουμε και να, ή να μην το δοκιμάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι η συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί δεν σχετίζεται με τη δημιουργία ενός δημόσιου ευρωπαϊκού οργανισμού που θα επιτελεί ένα γενικό καθολικό έργο όσον αφορά την έκδοση αξιολογήσεων, πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα ε, και κόστους. Το θέμα είναι ωστόσο ότι όσον αφορά την ε, αξιολόγηση των δημοσίων χρεών υπάρχουν ε, οι τεχνικές γνώσεις και η εμπειρία ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια αξιολόγηση βασισμένη στην τρέχουσα κατάσταση και στο έργο ορισμένων θεσμικών οργάνων της Ευρώπης. Εγώ πιστεύω ότι το να υποστηρίζουμε όπως ε, κάνει ο Ashley Fox ότι όλες οι χώρες θα είχαν τριπλό α σημαίνει σιωπηρά ότι οτιδήποτε κάνουμε σε αυτό το κοινοβούλιο και στους ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι περιττό. Διότι υπάρχει και το δημοσιονομικό σύμφωνο, το φυσκαλικό πακτό, όλα αυτά δηλαδή δεν ωφελούν σε τίποτα. Εάν όμως λοιπόν πούμε ότι οι οίκοι αξιολόγηση αξιολόγησης μπορούν να επιτέλουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, αλλά ε, όχι τα αυτόνομα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θεωρώ ότι αυτό δεν είναι πιστικό επιχείρημα. Επειδή επίση πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα σφάλματα που έχουν γίνει σε ορισμένε περιπτώσει αξιολόγηση εκ μέρου των οίκων τη αξιολόγηση. Δεν θέλω να δώσω ονόματα, αλλά μέχρι πριν από λίγο καιρό διάβαζα απόψεις και πολιτικού χαρακτήρα, όπως είπε ο κ. Λάμπερτς, στις οποίες αναφέρω, λέγανε ότι αν εσείς δεν κάνετε πολιτική λιτότητα θα σας υποβαθμίσουμε. Μετά από καμιά εβδομάδα οι αξιολογήσεις έλεγαν, με συγχωρείτε που το απλοποιώ τόσο πολύ, εάν δεν ε, εφαρμόσετε αναπτυξιακή πολιτική θα σας υποβαθμίσουμε. Αυτό πιστεύω θέτει το πρόβλημα της ισορροπίας και της πολυφωνίας απόψεων. Αυτού του τύπου την προβληματική πρέπει να μελετήσουμε και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε και αυτή την αξιολόγηση εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Ξέρω ότι το ζήτημα είναι φλέγον έχουν δίκιο όσοι λένε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει εντάσεις, αλλά στην πραγματικότητα οι εντάσεις υπάρχουν ήδη. Και αναρωτιέμαι μήπως αυτή εδώ είναι η κατάλληλη στιγμή και μήπως είναι σκόπιμο να έχουμε και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αυτή την πολυμορφία απόψεων και αυτά τα benchmark για τα οποία μίλησαμε που θα μπορούσαν να αφορούν την υιοθέτηση και την υλοποίηση ε, διαφορών κριτηρίων. Δεν θέλω να μακρηγορήσω υπερβολικά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε και να εμβαθύνουμε το ζήτημα της εναλλαγής. Αντιλαμβάνομαι τους ενδιασμούς του Βολφ Κλίντς, για παράδειγμα. Από φιλοσοφική άποψη θα μπορούσαμε ε, να το να αναφερθούμε σε αυτό ως ετερογενείς ε, σκοπούς ε προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα στόχο επιτυγχάνοντας το αντίθετο. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε την αναλλαγή αλλά όχι σταθεροποιώντας το λιγοπόλιο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την παρατήρηση αλλά θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι ούτως ή άλλως χρειαζόμαστε κανόνες και μέτρα με αυτό το κανονιστικό πλαίσιο που θα διατηρήσουν σταθερή την αρχή της μέγι, του μέγιστου ανοίγματο της αγοράς και του μέγιστου ανταγωνισμού στην αγορά των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Στην εισαγωγή μου είχα αναφέρει όλα τα σημεία στην τροπολογία για την tender procedure καθώς και τις παρατηρήσεις του Wolf klinz Ας τα μελετήσουμε όλα αυτά έτσι ώστε ξεπερνώντας την υπερβολική πολυπλοκότητα του μηχανισμού προτείνει η Κομισιόν να διατηρήσουμε ωστόσο αυτή την αρχή του ανοίγματο στον ανταγωνισμό, του μέγιστου ανταγωνισμού και της δυνατότητας άρσης των φραγμών εισόδου νέων ε, φορέων στην αγορά επιστολιπτικής αξιολόγησης. Εγώ πιστεύω και κάποια, ότι και κάποια άλλη σημεία που υπενθυμίσατε εδώ μας βρίσκουν σύμφωνους. Ε, λογικά όσα είπε ο κύριος Σιμών, ο Πίτερ Σίμων, για την ανάγκη καλύτερου επανακαθορισμού της πτυχής που σχετίζεται με τη σύγκρουση συμφερόντων. Έχω εμπιστοσύνη για αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να συγκλίνουμε αποτελεσματικά. Τέλος, πιστεύω, και αυτές είναι οι δύο τελευταίες μου παρατηρήσεις, ότι θα ήταν σωστό να εργαστούμε, όπως είχα προτείνει και εγώ εξάλλου, για την αστική ευθύνη υπό τους όρους που προτείνονται από τον κύριο Γκόζες, ώστε να μπορέσουμε και εδώ να διαφυλάξουμε την αρχή καθορίζοντας ωστόσο με καλύτερες και περισσότερες λεπτομέρειες ε, ένα κομμάτι του περιεχομένου και ορισμένες από τις αρχές. Και επίσης, όσον αφορά το ζήτημα των τρίτων χωρών, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε αναφορά όπως υπογράμμισαν οι Κλίντς και Γκοζές ε, σε όσα ε, κατέδειξαν ήδη και έχουμε διαπιστώσει ήδη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί χωρίς απαραίτητα να ανοίγουμε ξανά μια γενική συζήτηση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που για τα σχόλιά τους. Ε, εύχομαι ότι στις επόμενες συνεδριάσεις θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα βήματα προς τα μπρος και φυσικά θα αρχίσουμε να ε, εργαζόμαστε βάσει αρχικών υποθέσεων συμβιβασμού ώστε να μπορέσουμε αποτελεσματικά να ανταποκριθούμε στην πολιτική ευαισθησία και στην κοινή γνώμη όσον αφορά τους οίκους πολιτικες κανότητας την παρούσα Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους παρόντες. 7 Ιουνίου είπαμε θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας ώστε να ψηφιστεί η έκθεση αυτή και στην ε, Ολομέλεια του Ιουλίου. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι τελειώσαμε για σήμερα το πρωί. Σας αναμένω και πάλι στις 3 στην αίθουσα. Ευχαριστώ.